Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης ε, είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Αν όχι, εγκρίνονται τα πρακτικά.